Και συνάδελφοι, ξεκινάμε από την κατάσταση ή στην Μεσόγειο, διότι χρειάζεται να υπάρχει μια σφαιρική, συνολική, πολιστική προσέγγιση. Έχουμε τώρα το σχεδόν του και θα πρέπει όμω να σα αναφέρω ότι μία από αυτέ αναφέρει ότι ε, από τις 7 λεπτά μέχρι τις 8.30 οι, οι στέλνει. δεν πάει σε ξέρετε είναι Ελλάδα στο 7,5 με 9 είναι 7 με 8,5 ώρα. Οπότε έχουν το σχέδιο τη εκθέσεω και ευχαριστούμε του ε, ε, συντάκτα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο και έχουμε επομένω μόνο μία μισή ώρα. Σα φαίνεται πολύ, αλλά για κάτι τόσο σημαντικό δεν είναι τίποτα. Πρώτη για μια έκθεση για την οποία η καταληκτική ημερομηνία είναι η 8η Φεβρουαρίου, δεν είναι και πολλή χρόνο ε, για να έχουμε μία πλήρη έκθεση Οπότε σε αυτή τη μια μισή ώρα θα σας πω πόση ώρα θα μιλήσει ο καθένας και γι' αυτό συνάδελφοι θέλω να είσαστε συγκεκριμένοι και επίσης και οι πρόκειται να κάνουν τις εισηγήσεις τους και στα πλαίσια της εκθέσεως ιδίας πρωτοβουλίας πρόκειται να προχωρήσουμε σε αυτή την παρουσίαση πρώτα πρώτα από τους ε, συντονιστές και κατόπιν θα ακούσουμε τον κύριο Σάγκη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο την Home και Ιστορικών Υποθέσεων. Μετά θα έχουμε τον αναπληρωτή διευθυντή της ε, για Μετανάστευση, Δικαιοσύνη και Ασφάλεια, κατόπιν ο κ. Ντάνιελ Ντάιμ ο οποίος πριν από το, από το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντζα στη Γερμανία. Τον κάλεσαν οι συνεισηγητές και του είπα δύο κομμένε πριν τη συνεδρίαση και μου είπε ότι όλα αυτά τα συζήτησε με τους Και μια που δεν έχουμε τόσο χρόνο, θα ξεκινήσουμε ευθύ αμέσω την συζήτηση με τους δύο εισηγητές. Και ξεκινώ. Θα δώσω το λόγο πρώτα για να μας αναπτύξει τα βασικά σημεία του κειμένου στην Ρομπέρτα Μετσόλα. Ε, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και θα είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη και ευσύνοπτη αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα τεχνικό από ό,τι φαίνεται δεν είναι εκτός μικροφώνου τώρα. Okay, so, um, just say a few words and just... Δύο λόγια λέει ο πρόεδρος. να... Α, να πούμε τώρα μια δοκιμή για να δούμε αν παντού ε, λειτουργούν τα ακουστικά και αν ακούτε τους διερμηνείς όλοι. Όλες τις γλώσσες που έχουμε. Ακούνε όλοι τώρα την μετάφραση από τους διερμηνείς. έχουμε βεβαίως γερμανικά σήμερα. But it includes German, no? Just checking again, colleagues. Test, test. Όλοι ακούτε. Ακούτε τώρα. Όχι. Α, τώρα λειτουργεί. Μεταφράζεται προς τα γερμανικά αυτό το βιολό και το ακούτε. Το ακούτε. Ah, okay. Um, it does also say I should, I should, uh, could I just say, colleagues, my, my Συνάδελφοι, συμπαθάτε με εγώ, έκανα λάθο. Πάντως, δεν σας είπα ότι έχουμε και ε, μαλτεζικά, παθητικά και γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, σουηδικά, ουγγρικά, πολωνικά, σλοβακικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Οπότε, Ρομπέρτα, έλεγα ότι σου έδωσα το λόγο για να κάνεις την παρουσίασή σου. Πρέπει να με περιορίσω όμως, ε, πρόεδρε, για να σας πω τι έχει γίνει. Έχουμε αυτή την έκθεση που είναι 27 σελίδες και ε, ε, έγινε η του κειμένη πριν από λίγο για να το μελετήσουμε. τα Και είπαμε ότι θέλουμε να κάνει κάτι η για το μεταναστευτικό. Και όταν λέμε ότι πρέπει να γίνει αυτή η προσέγγιση δικομετικά ούτω ή αυτό ήταν ξέρουμε θα είναι δύσκολο, αλλά δεν ξέραμε ότι ε, δικομητικά λαϊκιστέ σε όλη την Ευρώπη και επίση μα ε, εμπόδισαν τα θέματα ασφαλεία, τα οποία εντοπίζει η Ευρωπαϊκή Πύρο. Οπότε δεν ήταν εύκολο το έργο μα. Ε, ε, Βεβαίω και εδώ που έχουμε συνηθίσει ο καθένα να τα λέει από το ιδεολογικό του μετερίζει, αλλά εάν θέλουμε να υπάρχει κάποια πιθανότητα κάτι συγκεκριμένο να περάσει, τότε όλοι ξέρουν ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη μικροπολιτική και να έχουμε μια τέτοια σφαιρική, συνολική προσέγγιση, ολιστική. Αυτό που θέλουν οι πολίτε. Οπότε ευχαριστώ την κυρία Κιέγγε, την συνεισηγήτρια, αλλά και όλου του άλλου που μα μίλησαν και που μα βοήθησαν. Και ξέρουμε ότι οι μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν στο μεταναστευτικό, οπότε και θα πρέπει να δούμε το, το κάθε μικρό σημείο και το τόσο ώστε να μπορέσουμε να βρούμε ένα γενικό ε, πλάνο και αυτό και προσπαθήσαμε να περιγράψουμε στην εκθεσή μας. Πρώτα πρώτα βλέπετε, στο γύρω στο κειμένου βλέπετε ότι η λέξη κλειδί είναι η αλληλεγγύη για οποιαδήποτε δράση που αφορά την μετανάστευση και αυτό θα πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε όλες μας τις ε, συζητήσεις και θα ξέρω ότι θα πρέπει να σα έχω στείλει πιο νωρί την έκθεση, αλλά είμαι σίγουρο ότι θα μπορέσετε να αναλύσετε ε, τι λεπτομέρειε τη επόμενε εβδομάδε επί τη βάση του εγγράφου εργασία, το οποίο ήδη συζητήσαμε στην Επιτροπή μα. Και τώρα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Να ξαναγίνουμε αυτά τα πράγματα περισσότερα, ούτω ώστε να σταματήσουμε ε, τον κόσμο από το να πνίγεται. Ε, και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις επιχειρήσεις διάσωση και είπαμε ότι η Frontex αλλά και το ναυτικό και επιχειρήσεις όπως η Σοφία έχουν ε, παίξει κάποιο ρόλο, έχουν σώσει ζωέ, αλλά θα πρέπει να προωθήσουμε και άλλο. Επίση τονίζουμε ότι όποιο βοηθάει ε, δεν θα πρέπει να κατηγορείται και να παραβαίνει στην ποινική δικαιοσύνη και για την Frontex. Είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε ε, ε τώρα και καινούργιε υπηρεσίε όπω την ακτοφυλακή να την αντικαταστήσουμε και είπαμε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση στα εξωτερικά σύνορα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε την μετανάστευση και επίσης να μπορέσουμε να έχουμε και εσωτερική ασφάλεια. Οποιαδήποτε ολιστική προσέγγιση σε αυτό θα πρέπει να έχει ως ε, σκοπό στο να αναχαιτήσουμε τους ε, εγκληματίες και τα δίκτυα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό έχει σημασία και όσον αφορά και τις ε, χρηματοοικονομικές έρευνες ε, τα οικονομικά τους, τις, τις κατασχέσεις που είναι σε προϊόντα εγκλήματος και είπαμε ότι θα πρέπει όσον αφορά την μετεγκατάσταση, αν είμαστε ένωση αξιών, ε, θα πρέπει να έχουμε και κοινή ευθύνη και υπευθυνότητα και θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να παίξει το ρόλο του. Οπότε αυτά τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τη μετεγκατάσταση είναι η σωστή κατεύθυνση. Αλλά μέχρι τώρα ποσοτικά δεν τα έχουμε πάει καλά. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους, ό,τι δεσμεύτηκαν και αυτό το κάνουν όσο γίνεται πιο σύντομα. Γιατί με την κατάσταση τώρα σε σχέση με το ότι έχουμε τώρα αυτέ τι ροέ χωρί προηγούμενο. Συνεχίζουν, έρχονται στα σύνορά μα και άρα ξέρουμε ότι χρειάζεται να υπάρχει μια νομοθεσία δεσμευτική. για με την κατάσταση ακριβώ όπω είπε και στο λογιών τη Κομισιόν για την μετανάστευση τώρα. Ε, θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε διατάξει για την προστασία του κόσμου και να έχουμε και κάποιο είδου ε, θεωρήσει διαβατηρίων ε, και κάποιους κανόνες για την ε, υποδοχή εάν θέλουμε να σταματήσουμε να τους εμπνευνούνται οι διακινητές και να βρίσκουν το θάνατο στα σύνορά μας. Τώρα αφορά τα σύνορα θα πρέπει να σταματήσουν οι, έλεγχοι ε, να ισχύει το, το, το Σέγγεν και να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Αυτό είναι προπόθεση για να μπορεί να λειτουργήσει σωστά το Σέγγεν και οπότε θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει αυτό το κοινό σύστημα ευρωπαϊκού ασύλου και να αντιμετωπίσει ότι υπάρχει και επίσης να ε, υπερασπίσει την ασφάλεια και την αρχή της ελεύθερης διακίνησης. Όλοι θα πρέπει να είναι ασφαλείς σε Βερολίνο, ε, Ρώμη, Βαλέτα, παντού. Και επίσης ε, υπάρχουν κάποιοι φόβοι λόγω αυτών των ροών, άρα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις του εξωτερικά σύνορα, εάν θέλουμε αυτοί οι φόβοι να διασκεδαστούν. Και όσον αφορά τώρα την κοινωνική ένταξη, ε, λέμε ότι είναι δυτή εδώ η διαδικασία και βέβαια είναι αυτό αυτονόητο ότι αυτοί που έχουν προστασία θα πρέπει να ε, έχουν ό,τι δικαιώματα δικαιούνται, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερο, ώστε οι οικογένειε να είναι ενωμένε και ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός των αξιών θεμελίων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε τώρα για το σύστημα του Δουβλίνου που από λεπτομέρειε και για όλα αυτά θα πρέπει να πούμε ότι σίγουρα δεν έχει πετύχει τους στόχους και ε, λέμε τώρα τι μπορεί να γίνει και τι πρέπει να συζητηθεί. Ξέρετε, δεν είναι όλοι επιλέξιμοι, δεν δικαιούνται όλοι προστασία όσοι έρχονται εδώ. Οπότε θέλουμε να υπάρχει επιστροφή ε, όσων δεν δικαιούνται προστασία. Μόνο 36 90% των όσων στείλαμε πίσω, αυτοί πραγματικά έφυγαν το 2014. Άρα θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί όσον το σύστημα επαναπατρισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα αυτό οπωσδήποτε θα πρέπει να γίνει. Και ή χαιρετίζουμε τον κατάλογο των ασφαλών χωρών τη Κομισιόν και αν θέλουμε να είναι αυτό ο κατάλογο υπουργείων για τα κρατημέλη, αυτό θα είναι ένα εργαλείο πάρα πολύ χρήσιμο για τη διαδικασία του ασύλου αλλά και τη του επαναπατρισμού. Τώρα, όσον αφορά τα hot spots, τα κέντρα καταγραφής των μεταναστών θα πρέπει να έχουμε ενεργά τέτοια κέντρα ε, και επίσης εδώ πέρα εξηγούμε τι θέλουμε ότι θα πρέπει να γίνει ούτως ώστε να βρούμε τις ε, αιτίες της μετανάστευσης και καταλαβαίνουμε ότι μακροπρόθεσμα θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο για τα γεωπολιτικά θέματα τα οποία ε, είναι οι αιτίες δηλαδή πόλεμος, φτώχεια, διαφθορά, έλλειψη ευκαιριών και όλος αυτός ο κόσμος αναγκάζεται ε, να μεταναστεύσει. Και αυτό θα αλλάξει μόνο αν εμείς βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να ανασυγκροτηθούν, όπως θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διαθέσουν τους πόρους ώστε να βοηθούν αυτές οι χώρες. Να βελτιώσουμε τις επενδύσεις, να βοηθήσουμε στην παιδεία, την εκπαίδευση και θα πρέπει το σύστημα του ασύλου να βελτιωθεί, να υπάρξει καλύτερη διαχείριση, ε, δικαιοσύνη επίση να βοηθήσει αυτέ τι χώρε και λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσει τι χώρε ούτω ώστε να έχουν ένα σύστημα ασύλου και να υπάρχουν ε, στατικές ένταξεις για να υπάρχει διεθνής προστασία. Ε, επίσης εδώ αναφέρουμε ε, το τελευταίο σχέδιο Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία. Και είπαμε ότι όλε οι πλευρέ θα πρέπει να τηρήσουν τα συμπεφωνημένα. Και η Τουρκία θα πρέπει να τηρήσει τι δεσμεύσει τη, ώστε να σταματήσει την λάθρο από Προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την χρηματοδότηση, θέλουμε τα πράγματα να έχουν περισσότερη διαφάνεια, να είναι πιο εύκολα και θέλουμε περισσότερε οργανώσει να μπορούν να εκμεταλλευτούν του πόρου που διατίθεται εκεί. γι' αυτό και είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το Emergency Trust Fund για την Αφρική και τα 1,8 δι τα οποία διατέθηκαν για αυτό το Ταμείο για την Αφρική. Θέλουμε στα κρατημέρια να συνεχίσουν να βοηθάνε Τώρα, όσον αφορά τι επιλογέ για την νόμιμη μεταναστεύση, τότε τα δικαιώματα των κρατομελών για να καθορίσουν το πόσο θα υποδέχονται από τι τρίτε χώρε που θέλουν κάποια δουλειά, αυτό είναι σαφέ. Όμως θα πρέπει τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να δούνε ε, τι και να παράγουν στην αγορά, τα οποία θα μπορούσαν να τα γεμίσουν αυτοί ε, από τις τρίτες χώρες. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει, πώς θα αναθεωρηθεί και πώς θα είναι η αναθεώρηση της οδηγίας για την μπλε κάρτα πιο φιλόδοξη, οπότε θα πρέπει να ε, καταπολεμήσουμε κάποιους ε, εργοδότες που τους πιο ευάλωτους τους ε, εκμεταλλεύονται και επομένω θα πρέπει να ξεριζώσουμε την εκμετάλλευση και επίση να στείλουμε στη δικαιοσύνη όλου εκείνου που εκμεταλλεύονται αντί να προστατεύουν τα θύματα. Επομένω, εδώ έχουμε μια μακροσκελή εντελεχή έκθεση αλλά είμαι ε, βέβαια ότι μπορούμε να την έχουμε σαν αφέτη εργασία. Ε, άλλα τέσσερα παιδιά από ό,τι γνωρίζουμε πνίγηκαν το Σαββατοκύριακο πριν καν μπορέσουν να μπουν στην Ευρώπη και θα πρέπει να δούμε ε, πώς θα σταματήσουμε όλες αυτές τις χιλιάδες ε, από όλους αυτούς που χάθηκαν μαζί με τα όνειρά τους άρα να διαχειριστούμε καλύτερα την ε, μετανάστευση και η αδιαφορία δεν είναι επιλογή και εναλλακτική. Ευχαριστώ Ρομπέρτα. Ε, τώρα θα πάρει το λόγο η Σεσίλ και η συνεισηγητρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από ένα χρόνο ε, το Κοινοβούλιο αποφάσισε να δώσει μια άλλη απάντηση ε, στο μεταναστευτικό ε, και αντί για την επίγουσα συνήθεια διαδικασία να ακολουθήσει μια διαφορετική ολιστική σφαιρική προσέγγιση. Ε, και γεννήθηκε επομένω αυτό το σχέδιο έκθεσης. Όπως η συνάδελφο Ρομπέρτα Μετσόλα υπογράμμισε ήδη, η εργασία αυτή αποτελεί μια σύνθεση των θέσεων των κύριων πολιτικών ομάδων και επομένω ε, αποτελεί και μια, έναν συμβιβασμό ε, πάνω σε συγκλίνουσες θέσεις που αποτελούν το κεντρικό σχήμα αυτής της έκθεσης. Ε, η Ρομπέρτα Μετσόλα ήταν ε, πάντα στη διαθέσιμη για συνεργασία ε, και χαίρομαι που ε, είναι ε, και χαίρομαι για την εργασία που κάναμε. Ε, σήμερα γίνεται 37 χρονών και συμφωνώ με όλα αυτά που είπε. Οι πολιτικές μας ομάδες δούλευσαν και γι' αυτό και θέλω να τις ευχαριστήσω και θέλω να ευχαριστήσω και την γραμματεία της ΛΥΜΠΕ για την διοικητική έτσι, υποστήριξη που μας έδωσε. Πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε, να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα κοινό κείμενο το οποίο αφορά και προτείνει ε, διάφορες προτάσεις παρέμβασης ε, σε διάφορα θέματα. Όπως θα διαπιστώσετε, ε, τα περιεχόμενα των διαφόρων, των διαφόρων εγγράφων εργασίας έχουν ενσωματωθεί εδώ. Αναφέρεται ας πούμε ότι το μεταναστευτικό φαινόμενο δεν είναι ένα φαινόμενο στο οποίο θα πρέπει να αντιταχθούμε αλλά θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίσουμε με ένα καλό ε, μείγμα ε, πολιτικής εσωτερικής και εξωτερικής. Επίσης ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί μακροπρόθεσμα έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι επίγουσες ανθρωπιστικές καταστάσεις καθώς επίσης και οι ρίζες, οι, οποίες, οι ρίζες του φαινομένου που βρίσκονται σε άλλες χώρες. Δεν θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να παραμείνουμε σε σε έναν αφηρημένο, σε ένα αφηρημένο επίπεδο αλλά θα πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο ε, μπορούμε με συγκεκριμένο τρόπο να ε, αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό. Νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχθεί τον πλήρως από τη δική μας πλευρά ε, όλες οι διαδικασίες διάσωσης. Ωστόσο, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να ε, βρουν έναν μόνιμο ευρωπαϊκό ε, μηχανισμό διάσωσης και με τρόπο ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο πλέον οι ζωές των, μετα, των προσφύγων. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα μετά από τη διάσωση να τους δώσουμε στους πρόσφυγες αυτούς ε, ε, και ε, μια ανθρώπινη αντιμετώπιση και την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να φτιάξουν τη ζωή τους. Ο μηχανισμός της διανομής θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικός και να δίνει την δυνατότητα στο μέτρο του δυνατού να λαμβάνονται υπόψη και οι επιθυμίες των προσφύγων όσον αφορά τον τρόπο, τόπο προορισμού τους αλλά έναν δεσμευτικό και μόνιμο μηχανισμό σημαντικού αριθμού των ετούντων άσυλο στο εσωτερικό των κρατών μελών, χωρίς όμως να παραβλέψουμε και άλλα στοιχεία όπως ας πούμε οι ανθρωπιστικές ε, επιχειρήσεις. Ε, η σωστή διαχείριση και η λογική διαχείριση ε, του προσφυγικού ζητήματος λύνεται και περνάει και μέσα από τη δημιουργία νόμιμων ασφαλών διόδων και διάβλων. Θα πρέπει οπωσδήποτε να

Ε, δούμε και να αντιμετωπίσουμε τις ε, πολλές δημοκρατικές προκλήσεις καθώς επίσης και την μεγάλη πρόκληση ε, των ανειδίκευτων εργαζομένων και με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται κάποιους γενικούς μηχανισμούς όσον αφορά τους προερχόμενους από τρίτες χώρες. Πάντα όσον αφορά τα οικονομικά στοιχεία. Εμείς καταδικάζουμε ε, με ε, επίταση οποιαδήποτε παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων και οποιαδήποτε κατάχρηση ε, των μεταναστών σε θέσεις εργασίας και υπενθυμίζουμε επίσης και όλα τα μέτρα τα οποία έχουν ήδη βάσει του κανονισμού 52 θεσπιστεί για τους εργοδότες που χρόνο των ε, ε, εργαζομένων και που δεν εφαρμόζουν τα ε, δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Οπωσδήποτε θα πρέπει να καθοριστούν οι ανάγκες οι εργασιακές στις αγορές των κρατών μελών και ε, με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουν να προωθηθούν αντιστοίχως ε, και οι πρόσφυγες. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε ε, μέτρα φιλόδοξα που κυρίως και εμπρότης να αφορούν την ε, ενσωμάτωση των προσφύγων και ε, κατά δεύτερον την ελεύθερη κυκλοφορία των προσφύγων. Πιστεύω ότι η μεγάλη πρόκληση είναι η κοινή μεταναστευτική πολιτική. Δηλαδή η μεγάλη πρόκλησή μας είναι να έχουμε πολιτική η οποία θα έχει σαν πρώτο ε, στόχο την ενσωμάτωση των προσφύγων στον κοινωνικό, εργασιακό και αστικό ιστό των χωρών μας ε, και επομένως να ε, τους δίδονται τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις που θα είναι αντίστοιχες με αυτές των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλούμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν σωστά το άρθρο 15 της οδηγίας για την υποδοχή και να διασφαλίσουν την ε, πρόσβαση στην αγορά εργασίας ε, των ε, δικαιούχων εννέα μήνες μετά την υποβολή του αιτήματο. Αναλύσαμε το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου και επομένως θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις παρά την, και όσον αφορά την ενεργή και όσον αφορά την ανάλυση που θα πρέπει να γίνονται όσον αφορά τις διαδικασίες σε πρώτη ε, φάση αλλά και όσον αφορά την ε, ε, οικογενειακή επανένωση το κράτος της πρώτης υποδοχής παραμένει υπεύθυνο. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η αρχή της διακριτικής ενημέρωσης. Οι χώρες στις όχθες των οποίων, στα παράλια των οποίων φτάνουν χιλιάδες ε, οδη, ε, πρόσφυγων μας οδηγούν στην ανάγκη αναθεώρησης ε, του Δουβλίνου. Δηλαδή να προβλεφθεί ένα κεντρικό σύστημα ε, το οποίο θα ε, συνάδει με την αρχή της επικουρικότητας ε, και της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Με ένα σύστημα μέσω του οποίου θα ορίζονται κατόφλια για κάθε χώρα πάνω από την οποία καμία επανατοποθέτηση ή επαναπροώθηση δεν θα επιτρέπεται ή μη μόνον εάν έχει καλυφθεί το κατόφλι της κάθε χώρας. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ληφθούν μέτρα κατά του τράφικινγκ και κατά της εμπορίας ανθρώπων ε, έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να πάρουν το καθένα ξεχωριστά και όλο μαζί ε, όλα τα μέτρα. Επίσης ε, θα πρέπει να πάψουν να υφίστανται οι λόγοι που σπρώχνουν τους μετανάστες, τους πρόσφυγες να ξεκινούν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν ήδη εργαλεία διεθνού συνεργασίας αλλά που θα πρέπει να βελτιωθούν και να εφαρμοστούν καλύτερα καλύτερα λαμβάνοντας υπόψη όλους τους εμπλεκόμενους, να υπάρξουν περισσότερα ε, προγράμματα περιφερειακή συνεργασία. Όσον αφορά δε το δικαίωμα ασύλου, αυτό είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι αναγνωρισμένο ε, και ε, από διεθνείς συμφωνίες αλλά και από τις συμφωνίες Ευρωπαϊκής και τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε προσπάθεια απομάκρυνσης ανθρώπων που έχουν ετηθεί ασύλου θα πρέπει να καταδικάζεται και να απαγορεύεται όλες ε, οι προσπάθειες θα πρέπει να γίνονται με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, τελειώνοντας να πω ότι βεβαίως δεν θεωρώ ότι έχουμε βρει τις τελικές λύσεις ε, και αυτό καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να προσπαθήσουν. Παρόλα αυτά επιτρέψτε μου να είμαι αισιόδοξη. Ήδη η εργασία μας έχει αρχίσει να παίρνει μορφή και διαπιστώνουμε από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι υπάρχει η βούληση αντιμετώπισης των αιτίων και των καταστάσεων καταστάσεων που οδηγούν ε, στο προσφυγικό. Ευχαριστώ. Και οι δύο σας ε, είπατε τι θέλετε να γίνει από πλευρά ε, Επιτροπής. Γι' αυτό η Επιτροπή και οι εξωτερικοί πάνελιστ θα μας πούν τι άποψη έχουν. Ξέρω ότι θα μπορούσατε να πείτε πολύ περισσότερα. Είναι η πρώτη φορά που αντικρίζουμε το σχέδιο αυτό και θα θέλαμε να αρκεστείτε στα 5-6 λεπτά. Σύγκεν από την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, διότι συμμετείχα και σε ε, ορισμένες ακροάσεις σας. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τις κυρίες ε, Μετσόλα και Κιέγγε για την παρουσίαση του σχέδιου έκθεσης ως προς την ε, κατάσταση στη Μεσόγειο και την ανάγκη μιας ολιστικής ε, προσέγγισης στο θέμα της μετανάστευσης. Τρεις είναι οι λόγοι. Καταρχήν η μεθοδολογία σας και η προετοιμασία της έκθεσης στη ΛΥΜΠΕ ήταν μια πολύπλοκη συνεργασία με εμπειρογνώμονες, με πολιτικούς, με ακαδημαϊκούς και υποβλήθηκαν πολλά έγγραφα εργασίας πριν από την τελική έκθεση. Είναι λοιπόν πολύ ε, σταθερό αυτό το πλαίσιο έτσι ώστε να κατανοήσουμε τις διάφορες συνιστώσεις της ΜΕΤΣ. Προετοιμάζοντας αυτή την έκθεση μιλήσαμε για αξίες και πολιτικές. Τις αποτιμήσατε. Πρόκειται για μια εκτενή έκθεση. Δεν αφορά μόνο την ολιστική προσέγγιση, αλλά καλύπτει και όλους τους τομείς που είναι σημαντικοί για τη μετανάστευση. Άρα εκφράζεται και τη στρατηγική σας άποψη ε, καταδεικνύοντας ότι δεν υπάρχει ένα κλειδί, ένα ενιαίο κλειδί για να αντιμετωπίσουμε την ε, μετανάστευση, αλλά ένα φάσμα μέτρων. Την έκθεση αυτή, μία έκθεση είχατε υποβάλει και τον Δεκέμβριο του 2014. Τώρα βρισκόμαστε στον Ιανουάριο του 2016. Είδαμε πως άλλαξε το φαινόμενο της μετανάστευσης, μας προσπέρασαν τα γεγονότα γιατί είχατε τη δυνατότητα δυναμικά να αποτιμήσετε και αναπτύξετε την στρατηγική σας άποψη. Ο πρόεδρος Γιούνκερ μίλησε για τη μετανάστευση ως πρώτη προτεραιότητα. Στη συνέχεια όμως για τα ε, νέα προγράμματα εργασίας ιδιαίτερα της Κομισιόν του 2016, είδαμε ότι υπάρχουν πολλές προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου. Και το πρόγραμμα εργασίας του 2016 έχει ένα συγκεκριμένο τίτλο. Δεν υπάρχει χρόνος για να συνεχίσουμε με την πολιτική business as usual. Είμαι σίγουρη ότι με την κοινή συζήτηση θα δώσουμε μια συνέχεια στην έκθεση και θα μας συνοδεύσετε για να μπορέσουμε όλοι μαζί να εγκρίνουμε τις ε, προτάσεις για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Γιατί η μετανάστευση θα παραμείνει θέμα πρώτης προτεραιότητας κατά τη θητεία σας και τη θητεία της Κομισιόν ξέρετε, το 2015 είχαμε πολλά ρεκόρ στις αιτήσει ε, χορήγησης ασύλου, 2 ε, εκατομμύρια και 1,8 ε, ως προς, τα περάσματα, ως προς το πέρασμα των συνόρων. Μιλήσαμε για τη λεκάνη της Μεσογείου από τον Ιούλιο-Αύγουστο σταθήκαμε σε ένα άλλο μέρος της ε, Μεσογείου, την Ανατολική Μεσόγειο και όχι την Κεντρική Μεσόγειο. Ως προς τις τάσεις που διαγράφονται είναι πολύ σχηδής γιατί αυξάνονται οι αριθμοί προσελεύσεων και θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στις χώρες έτσι ώστε να ληφθούν μέτρα και να μην δεχτούμε τα εσωτερικά σύνορα όπως έκαναν ορισμένε χώρες που στην ουσία ε, ανέγυραν φράκτες. Μιλάμε λοιπόν ε, για ένα πλαίσιο για την ε, μακροχρόνια πολιτική μας. Σε αυτή την ατζέντα της μετανάστευσης πολλές φορές στην Επιτροπή μίλησαμε για μέτρα αντιμετώπισης κρίσεων προσωρινών και μόνιμων, πιο μόνιμων. Προσπαθούμε να σταθούμε σε όλους τους πυλώνες όπως καλύπτονται από την έκθεσή σας. Θα πρέπει όμως να εστιάσουμε την προσοχή μας στη λειτουργία των πρώτων μέσων, δηλαδή να μην έχουμε διέλευση μεταναστών με μέσω παράνομων διάβλων. Βεβαίως τα χρήματα είναι πολύ σημαντικός παράγων, το αναφέρεται και η ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα μας δώσει νέα δημοσιονομικά μέσα για την εφαρμογή της ατζέντα. Ως προς το 2016 και τις προτεραιότητας μιλάμε για επανεγκατάσταση, hot spots, επιστροφές και σέγγεν καθώς και τα ευρωπαϊκά σύνορα και πρόταση ακτοφυλακής. Θα προτείνουμε και νέες προτάσεις για την αναθεώρηση του συστήματος ασύλου και ιδιαίτερα το σύστημα του Δουβλίνου για την νόμιμη μετανάστευση και επίσης θα πρέπει να δούμε και την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης μετά από τη Βαλέτα και τη Βουδαπέστη θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βρίσκουμε με αυτές τις διαδικασίες στο Ραμπάτ και στο Χαρτούμ. Η έκθεση αυτή είναι μια πολύ καλή συνεισφορά για τα επόμενα βήματά μας και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε αυτή την ατζέντα, για αυτή την ατζέντα για το μέλλον χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας με βάση τις προτάσεις σας για να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη μεταναστευτική κρίση που είχαμε μέχρι τούδε. Θα σταματήσω εδώ, δεν ήθελα να επεκταθώ. Ξέρω ότι είχατε πολύ περισσότερα να πείτε και μπορείτε να μας τα πείτε κάποια στιγμή, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και την άποψη των βουλευτών. Κύριε Ντία, σας καλωσορίζουμε ε, στην έκθεση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να συνοψίσετε κι εσείς τις απόψεις σας και θα ακούσουμε και τις απόψεις σας αργότερα. Ευχαριστώ. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση να είναι κανείς σύντομος για μια τέτοια έκθεση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι μεγάλη πρόκληση να είναι κανείς σύντομο σε μία έκθεση 27 σελίδων. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Το Συμβούλιο θα ήθελε να ευχαριστήσει και τις δύο συντάκτριες και θα ήθελα να ε, συγχαρώ και την κυρία Μετσόλα για τα γενέθλια της σήμερα. Η ολιστική προσέγγιση είναι σημείο κλειδί για να βρούμε ικανοποιητικές απαντήσεις. Δεχόμαστε το ψήφισμά σας της, του Δεκεμβρίου του 2014 ότι χρειαζόμαστε μια ολιστική προσέγγιση. Το Σέγγεν ε, υφίσταται πίεση με, και αυτό αφορά και το ευρύτερο και εκτιμένο. Για να παραμείνει το Σέγγεν θα πρέπει να γίνει πρόοδος σε θέματα της ε, δουλεμπορίας, της επαναφοράς και επιστροφής, καθώς και των hot spots. Επειδή η έκθεση ήταν διαθέσιμη δύο ώρες πριν από την συνεδρίαση, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο ε, δέχεται την ολιστική αυτή προσέγγιση, τη δική σας, που είναι εξαιρετική προσέγγιση ως προς την αλληλεγγύη. Η Προεδρία δέχεται ότι η αλληλεγγύη είναι η βάση του ευρωπαϊκού συστήματος. Χάθηκαν πολλοί ε, μετανάστες εξαιτίας των διακινητών. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την παράνομη διακίνηση. Είναι θέμα προτεραιότητας. Γι' αυτό την προηγούμενη εβδομάδα οργανώθηκε μία ε, διημερίδα στο Άμστερνταμ και το σχέδιο επαναπατρισμού και επανεγκατάστασης δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε με βάση τα hot spots και την προστασία των εξωτερικών συνόρων με την Frontex και το IASO. Θα πρέπει όμως να δημιουργηθούν περισσότερα hot spots στους επόμενους μήνες σε σχέση με την ανθρωπιστική ε, πτέρυγα συνιστόσα του ζητήματος το θέμα το έχει καλύψει ο κύριος ε, Λόπες Αγγιγιάρ, γιατί προσπαθούμε να δούμε και το καθεστώς της θεώρησης που θα δούμε από κοινού με τον συντάκτη. Ως προς την αναθεώρηση του Δουβλίνου, τον Μάρτιο θα υποβληθεί μία πρόταση και για το μηχανισμό του Δουβλίνου και για το θέμα του επανα ο Επίτροπος Αβραμόπουλος μας είπε ότι θα γίνει κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών με βάση και μία κλίδα κατανομή στα κράτη-μέλη. Το Συμβούλιο θα ήθελε αυτό το εξάμεινο να φτάσουμε σε μία πρόταση για τη σύνοριοφυλακή και την ακτοφυλακή. Θα προβούμε σε κοινέ προτάσεις με εσάς. Θεωρούμε όμως ότι και η Επιτροπή Παναπατρισμού είναι βασική συνιστόσα και τον Οκτώβριο πέρσι φτάσαμε σε συμπεράσματα. Η Ολλανδική Προεδρία θα προωθήσει αυτό το ζήτημα με τους επαναπατριζόμενους. Επίσης θα πρέπει να δούμε και τις ρίζες της κακοδεμανίας. Θα δώσουμε συνέχεια στις αποφάσεις της Βαλέτα και το πρόγραμμα της Τουρκίας καθώς και των Δυτικών Βαλκανίων. Θα πρέπει να βρούμε μία μακροχρόνια λύση. Προσπάθησα να μην ξεπεράσω τα πέντε λεπτά, τα κατάφερα σε τέσσερα. Yeah, spoke very fast. Μιλήσατε πολύ γρήγορα, λέει ο πρόεδρος. Sorry to rush you. Um, we've 10 or 11 uh, colleagues who wish to speak. Um, Τώρα αφήνετε χρόνο για τους αδελούς οι οποίοι θέλουν να μιλήσουν, αλλά μπορείτε να δευτερολογήσετε αργότερα. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα έχουμε κάποιον ε, προσκεκλημένο εκτός κοινοβουλίου ε, ένας ε, καθηγητής πανεπιστημιακός θα μιλήσει για πέντε λεπτά. Ξέρω ότι θα θέλετε να μιλήσετε περισσότερα, αλλά τι θέλετε, ένα διαδικαστικό, ναι. Γιατί για δεύτερη φορά δεν έχουμε εδώ ε, διερμηνείς από τα και προς τα τσεχικά έτσι το κοινοβούλιο δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά έγινε μια φορά αυτό και τώρα γίνεται και δεύτερη φορά που παραπονούμεθα το θέμα δεν είναι εδώ να ξέσκω τα αγγλικά μου το θέμα είναι να μιλούμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα και είναι δύσκολο δεν έχω το χρόνο να προετοιμαστώ. Βλέπω εδώ το μας και βλέπω ότι όντως δεν έχουμε ε, τσέχους διερμηνείς και όντως αυτή είναι η δεύτερη φορά. Οπότε αυτό θα το σημειώσω. Ε, δεν, είναι θέμα να δεν καταλαβαίνεις αγγλικά, αλλά θες να τα ακούσεις ε, στη γλώσσα σου. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, το κατανοώ, οπότε θα το δούμε. Γιατί έχουμε διάφορες γλώσσες που μας λείπουν σήμερα. Έχουμε όμως, ξέρετε, μόνο ένα θέμα. Είναι Στρασβούργο, είναι Δευτέρα, τέλος πάντων. Αυτό θα το κοιτάξουμε για να μην επαναληφθεί. Ευχαριστώ για αυτό το ευχαριστώ και τώρα δίνουμε το λόγο στον καθηγητή Τιμ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να σας ευχαριστήσω που με προσκαλέσατε. Μην είπατε ότι θα σας ε, παρουσιάσω μια άποψη κάποιου εξωτερικού, κάποιου πανεπιστημιακού. Πρώτα πρώτα να δούμε τα νομικά, μια που είμαι νομικός, Πολλές φορές έχουμε ε, διάφορα που λένε ότι αυτό είναι το σωστό. Να δούμε τι έγινε με τη σύμβαση της Γενέβης, τα δικαιώματα των ε, μεταναστών. Αυτό δεν το αμφισβητώ. Απλώς να σας τονίσω ότι από πλευράς νομικής είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να ε, βρει ακριβώς ποιες είναι οι συνέπειες ε, των πολιτικών που θέλετε να υιοθετούν γιατί η σύμφωση της Γενέβης είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Κανείς δεν θα πρέπει να επαναπατρίζεται εκεί που κινδυνεύει να διωχθεί. Και βέβαια πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι αυτή η απαγόρευση της επαναπρόθεσης δεν αποτελεί δικαίωμα του να διαλέξει κανείς τη χώρα εκεί όπου κανείς δεν έχει δίωξει αυτό φαίνεται αφηρημένο, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο κριτήριο για τέτοιες περιπτώσεις ροών. Εκεί που έχουμε τη συνθήκη της Γενέβης που λέει ότι μια ικανοποιητική λύση δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς διεθνή συνεργασία. Για να μην μακρηγορώ, η προστασία δεν χρειάζεται να την εγγυηθούμε για συγκεκριμένη χώρα. Θα πρέπει, όπως λέει η συνθήκη, να υπάρχει διεθνή συνεργασία. Και επίσης ε, δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία χωρίς να έχουμε διακρατικές συμφωνίες που να κατοχυρώνουν το δικαίωμα του να διαλέγει κάποιος που είναι ελεύθερος από διοξύ είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε αλλού. Και το Κοινοβούλιο επομένω συμμετέχει σε αυτή την συνεργασία, στις επιλογές και όλα αυτά βέβαια λαμβάνει υπόψη και τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί όλα αυτά καλεί ε, όλα αυτά λέει η συνθήκη της Γενέβης όταν πρέπει να γίνουν σεβαστά για τη συνεργασία. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα όρια ε, του κοινοδοτικού έργου. Όποιο έχει κοιτάξει την ολογία τη μεταναστευση, ξέρει ότι οι διασυνοριακέ κινήσει είναι περίπλοκα φαινόμενα και υπάρχουν πολλέ μεταβλητέ. Και οπότε αυτό το οποίο είναι σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια σφαιρική ολιστική προσέγγιση και θα πετύχει η πολιτική τη μεταναστευση μόνο αν δείτε όλες αυτές τις μεταβλητές των διεθνωριακών κινήσεων και ερών σε οποιαδήποτε γερμανική εφημερίδα μπορεί να διαβάσετε ότι σήμερα η κατάσταση δεν αφορά μόνο μακρόπινες λύσεις χρειάζονται και λύσεις βράχοι πρόθεσμες για να βρεθούν θα πρέπει να δοθούν κάποιες προτεραιότητες δεν είναι δυνατόν να έχετε σε λίγους μήνες την ολιστική προσέγγιση αλλά ποιε θα είναι οι προτεραιότητε, εσεί ε, είσαστε η αρχή του προπολογισμού, ε, και ασχολείστε με νομοθεσία και τα δημισιονομικά ε, και ακριβώ αυτό γίνεται πολλές φορές. Υπάρχει μια διαδικασία νομοθετική και ακολουθούν τα των ε, πόρων, της εκταμίας των πόρων. Και στην, στην Ευρώπη το θέμα είναι πώ θα εφαρμοστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο και για να έχετε πολιτική ασύλου θα πρέπει να δεχτείτε ότι πολλά τα προβλήματα δεν είναι δυνατόν να λυθούν μόνο από νομοθεσία και μόνο από την εκταμείωση των πόρων. Θα πρέπει να διευρυνθεί ε, ε, η Άσο και τη, ε, η εντολή και της Frontex ναι, έχετε αυτόν τον κατάλογο των ασφαλών χωρών και ίσως θα πρέπει να απλουστεύσετε τους τόσο περιπλοκούς κανόνες γιατί αυτό αποτελεί έναν φραγμό στην υλοποίηση του κεκτημένου. Βεβαίως και χρειάζεται νομοθετική δράση αλλά δεν είναι αυτό το πρώτο εργαλείο το οποίο θα, θα δώσει τις λύσεις στην κρίση. Βέβαια έχουμε και τον κανονισμό του Δουβλίνου. Αυτό είναι εξαίρεση. Ε, στην πρακτική είναι όλο ένα και πιο άσχετος και πάσχει από κάποιες αδυναμίες και αν θέλετε να βρείτε μια εναλλακτική τότε θα πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα ασύλου. Αυτό το οποίο μαζί με το Δουβλίνο πολλές φορές συμβαδίζει και έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδεθούν τα εσωτερικά συστήματα που μας αποτρέπουν από να έχουμε κοινό σύστημα. Άρα η συνθήκη ο κοινωνισμός του Δουβλίνου θα τεθεί να αμφιβόλως αργά ή γρήγορα. Θέλω να σας πω τώρα κατακλείδη ότι κάθε νομοθεσία για το σύστημα ασύλου είναι χτισμένη γύρω από έναν άξονα. Ο άξονα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχουν εξατομικευμένε διαδικασίε για τι ιδιομορφίε τη κάθε συγκεκριμένη περίπτωση επί τη βάση κάποιε ε, ακρόσει και κάποιου μηχανισμού περιπλοκού ενδίκων μέσων. Ε, και έχουμε φτιάξει αυτή την πολύπλοκη νομοθεσία πολλών εκατοντάδων σελίδων στην επίσημη εφημερίδα γύρω από αυτήν την εξατομικευμένη διαδικασία και για τους πρόσφυγες και για όσους χρειάζονται κάποια προστασία. Όμως θα πρέπει να δούμε το ότι αυτή η εξατομίκευση ε, πώς θα βοηθήσει όλες αυτές τις εισρωές οι διαδικασίες. Παίρνουν χρόνο. Χρειάζονται επίση ε, διοικητικές ε, ενέργειες, οπότε η διοικητική μηχανή βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση. Άρα με τη σημερινή κρίση ίσως θα έπρεπε να αναστείλουμε, να συμπληρώσουμε τουλάχιστον έστω και προσωρινά αυτή την εξατομίκευση και να έχουμε μια γενικευμένη διαδικασία σύμφωνα με κάποια οδηγία προστασίας και αυτά από νομοθετικής πλευράς ε, και βέβαια αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει βέβαια ε, μια συμφωνία για το πρόβλημα του κανονισμού του Δουβλίνου γιατί χωρίς αυτό δεν μπορεί να γίνει ε, καμία, κανένα βήμα και κυρίως να υπάρχει ε, κοινή ανάληψη των βαρών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δύσκολο θέμα και τώρα συνάδελφοι έχουμε 12 που έχουν ζητήσει το λόγο. Παρακαλώ πάρα πολύ, περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο και 8 Φεβρουαρίου λίγη προθεσμία των τροπολογιών. Ξεκινούμε με τους πιο συζητητές. Κύριε Στίβενς, έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις εισηγήτριες οι οποίες ανέφεραν ότι η διαδικασία είναι μακροπρόθεσμη. Πρέπει να σας πω ότι στην αρχή ε, στην σκέφτηκα ότι η έκθεση ε, είναι κάτι σαν χαμένη ευκαιρία. Δηλαδή όντως ε, καταγράφει μια σειρά στοιχείων και κάνει παρατηρήσεις. Αλλά αυτό που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση είναι η πραγματική βούληση να κάνουμε κάτι διαφορετικό και να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο. Λίγα στοιχεία είναι νέα σε αυτήν την έκθεση και λίγα είναι τα, ε, ε λίγες είναι εναλλακτικές προτάσεις. Στην ουσία επαναλαμβάνουμε τα ίδια, άρα δεν προχωράμε και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ήλπιζα να βρω και κάποιες ιδέες με τις οποίες θα μπορούσα να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω, αλλά να είναι νέες ιδέες. Ε, και δυστυχώς δεν είδα τίποτα τέτοιο. Ελπίζω πάντως ότι οι τροπολογίες και οι διαδικασίες ε, ε, συμβιβαστικών τροπολογιών θα δώσουν την δυνατότητα να προσθεθούν αξίες και νέα στοιχεία σαν Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είμαστε σαφείς σχετικά με το τι πραγματικά θέλουμε, σχετικά με το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα και πώς θα τα επιτύχουμε ε, τα νέα αυτά βήματα. Βεβαίως ε, κατανοούμε ότι με την ανάμειξη τόσων πολλών πολιτικών ομάδων ε, θα πρέπει να υπάρχει κάποια δημιουργικότητα. Αλλά, αλλά τώρα οι εκλογείς μας, οι πολίτες μας στρέφονται προς εμάς και περιμένουν να δουν τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να συζητήσουμε επίσης και την νόμιμη μετανάστευση. και θα θέλαμε αυτό να συμπεριληφθεί στη γενική συζήτηση για την ε, μετανάστευση. Επίσης, ε, οι ε, ικανότητες θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν μιλάμε για εργαζόμενους και φυσικά θα πρέπει να δούμε και το δημογραφικό πρόβλημα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες από τις οποίες προέρχονται. Ε, οι ε, μετανάστες. Τώρα, αυτά που αναφέρονται σχετικά με την αναθεώρηση του κώδικα των θεωρήσεων Visa Code ε, δεν νομίζω ότι μπορούν να απαντήσουν στους προβληματισμούς μας και την αλλαγή ας πούμε στο καθεστώς των μπλε θεωρήσεων. Νομίζω ότι με αυτές τις μπλε θεωρήσεις και με τις και, με, όσον αφορά αυτά που αναφέρονται για τις ποσοστώσεις νομίζω ότι δεν να κάνουμε και πολύ θαραλέα βήματα. Είναι σαν να μετακινούμε τα έπιπλα την ώρα που έχει πιάσει φωτιά το σπίτι. Ε, ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε για επαναπροωθήσεις εν θερμό, αλλά ε, θα πρέπει να δούμε κάποιες διαδικασίες επιστροφής, θα πρέπει να δούμε κάποιους τρόπους με τους οποίους να λειτουργήσουν καλύτερα όλες αυτές οι διαδικασίες. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα και να προστατέψουμε την περιοχή Σέγγεν. Αυτά είναι στοιχεία Βεβαίω, επί των οποίων μπορούμε να, συζητή, να συμφωνήσουμε όλοι το ζήτημα και το ζητούμενο μάλλον είναι με ποιο τρόπο θα τα συζητήσουμε, με ποιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε το σύστημα του Δουβλίνου. Ε, γιατί είδαμε ότι ε, πολλαπλώ δεν λειτουργεί, αλλά πώς θα το αλλάξουμε, πώς, προς ποια κατεύθυνση θέλουμε να το αλλάξουμε, πώ μπορούμε να βελτιώσουμε ε, την πρόταση του, του Δουβλίνου. Ωραία, θα αναθεωρηθεί. Θα πρέπει επομένως να ξεκινήσουμε να ψάχνουμε εναλλακτικές, αλλά για την ώρα δεν βλέπουμε τις εναλλακτικές στην έκθεση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν με τρίτες χώρες, αλλά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς ε, με τους εαυτούς μας. Ε, νομίζω ότι στις συμφωνίες με τις τρίτες χώρες τελικά ε, δεν, δεν κερδίζουμε τίποτα. Δηλαδή κάνουμε κάποιες κινήσεις, κάποιες προσπάθειες και τελικά εκείνες οι χώρες συνεχίζουν με το δικό τους τρόπο να λειτουργούν. Πάντως πρόκειται για μια έκθεση ε, η οποία, την οποία βρίσκω πάρα πολύ ε, ε, σημαντική. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να προκύψουν νέες ιδέες, νέες προτάσεις για να βοηθήσουμε να, και να συμβάλλουμε όλοι γιατί ώστε τα επόμενα χρόνια να έχουμε μια πολύ πιο καλή πολιτική ασύλου. Ξέρω ότι μακρηγόρησα αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει τουλάχιστον στη δικιά μας Επιτροπή να μπορέσουμε σε βάθος να συζητήσουμε τα θέματα Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε τώρα να συζητήσουμε σε βάθο. Έχουμε και άλλους συναδέλφους που προσθέθηκαν. Ε, τώρα ολοκληρώνεται, κλείνει ο κατάλογος των αγοριτών, αλλά ε, ήθελα να πω ότι στην έκθεση γίνεται λόγος για τα πάντα. Ε, ξέρω ότι δεν είχατε δει την έκθεση μέχρι τώρα, τη βλέπετε τώρα πρώτη φορά. Ε, και ε, μέσα σε δύο λεπτά πρέπει να πείτε όλα αυτά τα οποία ε, σας είναι ιδιαίτερος προσφυλή δεν είναι δυνατόν ξέρω ότι όλοι θέλουμε να συζητήσουμε για τα πάντα αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν και δεν θα είναι δυνατόν σε αυτή τουλάχιστον τη συνεδρίαση λοιπόν έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών από την ομάδα ALDE η κυρία Βίξτρομ Σκιώδης η Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Πρώτα απ' όλα θα ήθελα ε, να ε, δώσω τις ευχές μου στη Ρομπέρτα που έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Ε, δεν θα σου δώσω δώρο, αλλά δεν θα σε δυσκολέψω κιόλα. Θα σου πω συγχαρητήρια για τη δουλειά ε, που ε, έκανες. Ε, η άσκηση αυτή ήταν πρωτόγνωρη. Αυτή η ολιστική προσέγγιση ήταν διαφορετική, δεν είναι πάντα στο ραντεβού, αλλά παρόλα αυτά και δεν είναι πάντοτε παρούσα, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθεια έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι μπορούμε να ε, κάνουμε κάποιες ε, τροποποιήσεις ε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε λίγο αργότερα αυτή είναι την συνολική προσέγγιση που ζητάει η κυρία Στίβενς. Νομίζω ότι έχουμε ήδη αυτή την έκθεση αυτή και είναι σημαντικό που μπορούμε να την συζητήσουμε και αυτό είναι πολύ καλό. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την μετανάστευση σαν τέτοια, δηλαδή την νόμιμη μετανάστευση και την μετακίνηση, τη μετανάστευση των προσφύγων. Και χαίρομαι λοιπόν που και η νόμιμη μετανάστευση και τα περί αυτήν έχουν συμπεριληφθεί. Όπως ε, είπα, ε, μία ένωση μοιρασμένων ε, αξιών θα πρέπει να είναι και μία ένωση μοιρασμένων ευθυνών και εκεί έχουμε αποτύχει μέχρι τώρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει πλήρης αναμόρφωση του, της ηθίκης του Δουβλίνου γιατί έχει καταρρεύσει πλήρως και επομένως θα πρέπει να τροποποιηθεί. Ε, ε, η συνθήκη αυτή έγινε τον 20ο αιώνα, είμαστε πλέον στον 21ο και επομένως θα πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο στη διάθεσή μας το οποίο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις ε, νέες ανάγκες. Βεβαίως η ιστορική συνεργασία θα πρέπει οπωσδήποτε να προσθεθεί όχι μονάχα μεταξύ των κρατών μελών αλλά και ανάμεσα στις, ε, τις, ε, υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και τα κράτη-μέλη. Και επίσης όταν μιλάμε για μία ε, δίκαιη κατανομή, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια καλή αρχή, μια καλή άσκηση να συνεχίσουμε την προσπάθεια και ελπίζω ότι η Ρομπέρτα θα περάσει καλά το βράδυ των γενεθλίων της. Ναι, δεν θέλω να σας πιέζω, λέει ο Πρόεδρος, αλλά πρέπει. Ε, ας με αγνοήσετε αν δεν θέλετε να με λάβετε υπόψη σας. Η κυρία Σπινέλη παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τις δύο συντάκτριες για την εξαιρετική τους εργασία. Επειδή έλαβα αυτή την έκθεση αρκετά αργά, μπορώ να σας πω, ε, να κάνω ένα μερικό σχολιασμό. Είναι μια πολύ καλή βάση εκκίνησης. Υπάρχουν ε, στοιχεία που μπορούμε να εκτιμήσουμε. Θα πρέπει να έχουμε ένα ε, εύρωστο σύστημα διάσωσης, επίσης νόμιμες οδοί με βάση και το κανονισμό του 2001, επίσης η ανθρωπιστική διάβλη και ένας σωστός μηχανισμός εγκατάστασης. Βεβαίως υπάρχουν διαφορετικές μορφές ανθρωπιστικής βοήθειας, δεν θα πρέπει να υπάρξει ποινικοποίηση του όλου συστήματος. Όμως ε, δεν θεωρώ ότι το smuggling θα πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ε, συνοπτικά ως απόλυτα αρνητικό. Σε σχέση με την έλλειψη αλληλεγγύης μεταξύ κρατών μελών, εγώ θα επέβαλα πιο αυστηρές κυρώσεις κατά των κρατών μελών που δεν εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο ή δεν δέχονται να συνεργαστούμε βάση το άρθρο 80. Υπάρχουν ορισμένα σημεία που δεν με βρίσκουν καθόλου ως προς τον επαναπατρισμό, τη σχέση με τις τρίτες χώρες και ιδιαίτερα το θέμα της Τουρκίας, καθώς και τη τον κατάλογο των ε, σίγουρων σημείων επαναπατρισμού και των hot spots. Νομίζω ότι δεν κρίθηκαν σωστά μέχρι τώρα τα hot spots και τα είδαμε συνοπτικά. Από τους, από τους πράσινους κυρία Σαρτζεντίνη. Δεν ζήτησα το λόγο. Παρετούμε. Η FTD. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο. Ο κ. Φοντάνα από το ΙΕΝΕΦ. Ευχαριστώ. Εντάχει το έγγραφο θα πρέπει να το εμβαθύνουμε αρκετά και επιφυλασσόμαστε για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τις συντάκτριες διότι εργάστηκαν πολύ σκληρά. Αυτό ισχύει και για τους σκιώδεις. Υπάρχουν βεβαίως ε, στοιχεία που δεν μας πείθουν τόσο πολύ. Εμείς θα θέλαμε να είναι πιο σαφής η κατάσταση τη στιγμή που μιλάμε για επαναπατρισμό γιατί θεωρούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον επαναπατρισμό για αυτούς που δεν έχουν δικαίωμα χορήγησης ασύλου. Και θα θέλαμε κάτι το πιο συγκεκριμένο. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης και το γεγονός ότι ίσως χρειάζεται εργατικό δυναμικό, αλλά όχι σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Δεν είναι ίσα στις ανάγκες τους όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Γιατί έχουμε μετανάστες που βρίσκονται εδώ πολλά χρόνια και χάσαν την εργασία τους. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό, αλλά θα συνεισφέρουμε και εμείς ως προς τις τροπολογίες, έτσι ώστε το κείμενο αυτό να τύχει ευρύτερη συμφωνίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λόμπες Αγγίγιαρ. To make it short, so first, take... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλά, είναι δεδομένο ότι και εγώ, όπως όλοι θα συγχαρούμε την ε, Ρομπέτα και την ευχηθούμε και ε, βέβαια για το έργο και της Έλσινς για της κυρίας Κασέτου Κέγγε. χαιρετίζουν την προσπάθειά τους, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε να συνοψίσουμε τι πρέπει να προσθέσουμε στο κείμενο μέσω των τροπολογιών. Οπότε πέραν αυτής της ολιστικής, σφαιρικής και ενδελεχούς αναλύσεως όλων των μεταβλητών εδώ, ακόμη λείπει λείπει η επίκριση προς τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο που δεν μπόρεσαν να εφαρμόσουν τους δεσμευτικούς κανόνες δικαίου. Υπάρχει το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο. Δεν το εφήρμοσαν. Μιλούμε για τη μετεγκατάσταση, μιλούμε για όλα αυτά τα σχέδια και προγράμματα τα οποία το ίδιο το Συμβούλιο έχει αποφασίσει αλλά τελικά τα περισσότερα κατημέλη δεν τα ετήρησαν. Και βέβαια η προσφυγή στη διαδικασία επιπαραλήψης της Επιτροπής ακόμα είναι ε, ημιτελής. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και όσον αφορά το ενδιαφέρον του βιβλίου και όσον αφορά τις διαδικασίες για ανθρωπιστική προστασία και για το θέμα των ανθρωπιστικών θεωρήσεων διαβατηρίων Γιατί υπάρχουν ε, κανόνε που έχουμε στη διάθεσή μα. Ε, οι κανόνε όμω αυτοί πρώτα-πρώτα ε, δεν είναι ξεκάθαροι. Και επίση δεν είναι αποτελεσματικοί. Ακόμα και όταν εφαρμόζονται. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια αναθεώρηση. Θα πρέπει να ξαναδούμε αυτόν τον, αυτή την, την κωδικοποίηση των διατάξεων για την ανθρωπιστική θεώρηση διαβατήριου. Όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε με τις συνεισηγητρίες ακριβώς για να ανοίξουμε τον δρόμο ε, να ε, δοθούν λύσεις από νομικές, λύσεις που τώρα απουσιάζουν. Μα γι' αυτό ακριβώς που έχουμε τόσους ετούντες άσυλο, τόσους ε, πρόσφυγες που αναγκάζονται να ρισκάρουν τη ζωή τους ή τελικά να χάσουν και τη ζωή τους γιατί είναι απελπισμένοι ε, σε αυτή τους την προσπάθεια να χτυπήσουν την πόρτα της ε, Ευρώπης. Και φυσικά δεν είναι ο παράδεισος ε, αυτή η πόρτα όπως λέει το τραγούδι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κέρχοπ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τι συνηγητρίες. Βεβαίω και το δεύτερο ήταν δύσκολο, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσω με την Χέλγα Στίβεν, τη συνάδελφο. Είδα αυτό το θέμα για την ε, μόνιμη κατάσταση ε, αλλά δεν νομίζω θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας ε, στις προτιμήσεις του ετούντος, άσυλο για το πού θέλει να εγκατασταθεί. Από ό,τι ξέρω, η Ευρώπη είναι γεμάτη από ασφαλείς χώρες και όταν κανείς ε, προσπαθεί να σώσει τη ζωή του ε, και γίνεται πρόσφυγας ε, δεν είναι δυνατόν να του ικανοποιηθεί αναγκαστικά πρώτη του επιλογή. Θα πρέπει βέβαια να υπάρξει ένταξη στι κοινότητέ μας αυτών των ε, πρόσωπων. Θα πρέπει να δούμε τα παραδείγματα της αλληλεγγύη, είναι με τα σωστή κατεύθυνση και ήρθε την περσμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μας είπε ότι το σύστημα που εφαρμόζεται ε, χαρακτηρίζεται από έλλειψη ελεγγύης και άρα είναι αποτυχημένο. Δεν μπορεί όμως να επιβάλλει την ελεγγύη σε χώρες ή σε ηγέτες. Ε, θα πρέπει να υπάρχει στήριξη του εκλογικού σώματος. Και αυτό το οποίο δεν έχουμε είναι ένα σύστημα θα πρέπει να προσέξουμε τι γίνεται με τη μετακατάσταση, τι γίνεται με την υποπτία από την ε, Διεθνή Υπαδιαρμοστία των Σπουδίων Πρόσφυγες και επίσης λέει εδώ ότι θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις εθελούσιες στους επαναπατρισμούς. Εγώ ε, έχω σε μια άλλη κρίση χρηματίσει υπουργό και θέλω να σας πω ότι αυτή η μέθοδος δεν αποδίδει. Βέβαια η μικροπολιτική και οι συμβιβασμοί είναι φραγμόσιμη μια τέτοια έκθεση. Άρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και να είμαστε στους επόμενους μήνες πιο φιλόδοξοι. Κυρία Μουσολίνη, εκτός μικροφώνου. Εγώ σας ευχαριστώ συναδέλφοι για το έργο σας. Είναι περίπου αυτό το οποίο κάνατε γιατί έχουμε αυτό εδώ την πλατφόρμα που θα πρέπει να την είχατε σαν βάση δουλειά σε αυτή την προσέγγιση την ολιστική είναι κάτι το οποίο τώρα λείπει στην Ευρώπη μια τέτοια προσέγγιση όμως καταλήξατε σε ένα κείμενο που την υπόψη όλοι αυτούς τις δυναμικές μεταβλητές αυτά τα οποία συνέχεια μεταβάλλονται γιατί έχουμε τώρα αυτά τα τείχη που ορθώνονται από τα διάφορα κράτη. Είχαμε την ε, προσωρινή αναστολή του Σέγγεν ή ίσως και όχι τόσο προσωρινή αναστολή. Είναι περίπλοκη που είναι σε κατάσταση και γι' αυτό νομίζω ότι πρόκειται για μια προσέγγιση σημαντική, για μια έκθεση σημαντική, καλή αφετηρία και άκουσα τι είπε η συνάδελφος Κέγγε θα πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι σε μια τόσο τραγική κατάσταση όταν βλέπουμε ότι πρέπει, θα γίνουν όλα αυτά τα προγράμματα και είπαμε θα, θα πρέπει να βρεθεί δουλειά σε 9 μήνες και τι θα γίνει με τον γενικό ιστό στην ε, Ιταλία. Καλά και εγώ πρέπει ότι μετανάστες. Δηλαδή βλέπουμε ότι όλο το πρόγραμμα για τους νέους δεν επέδωσε ούτε μια θέση εργασίας για αυτούς. Επομένως θα πρέπει να ξαναδούμε αυτές τις σωστές πρωτοβουλίες. Τι θα γίνει με τον κοινωνικό ιστό, πού θα κολλήσουν αυτά. Και εμείς ως ε, συνιστόσα για την προσωπία θέλουμε ένα τέλειο κείμενο και οπότε θέλουμε για τις ροές να υποβάλουμε κάποιες ε, τροπολογίες. Επίσης άκουσα τον κύριο τον καθηγητή τον κύριο Τιμ που μας είπε για την δυνατότητα του να ε, έχουμε κάποια διαφορετική προσέγγιση έστω και για λίγο από την γενικευμένη από την περιπτωσιολογική σε μια γενικευμένη προσέγγιση. Πολύ σημαντικό αυτό και θα πρέπει να δούμε τι πρότυπα θα έχουμε. Πώς είναι να έχουμε μια ομοιομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια τέτοια κατάσταση όπου η κάθε χώρα προσπαθεί να ανέβρει λύσεις για μια τέτοια κατάσταση κατεπίγουσα. Οπότε δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με αυτή την πρόταση. Πρέπει να το κάνουμε, να το εφαρμόσουμε αυτό. Υπάρχουν περισσότερες πρωτοβουλίες για την μετανάστευση. και να υποβάλουμε και τις τοπολογίες για τις ροές αυτές και να εξετάσουμε και το θέμα ότι οι περισσότεροι είναι άντρες και πάρα πολύ λίγες οι γυναίκες. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, επανειλημμένα ε, ακούσαμε σήμερα να γίνεται λόγος για μετανάστευση, νόμιμη μετανάστευση, πρόσφυγες, προσφυγικό κτλ. Όλα αυτά είναι φλέγοντα ζητήματα. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω τις δύο εισηγήτριε οι οποίες ανέλαβαν δύσκολο έργο και νομίζω ότι με την έκθεση τους οι δύο συνάδελφοι δείχνουν ότι εάν πραγματικά θέλουμε να έχουμε καλές πολιτικές σε αυτό το τομέα ε, δεν μπορούμε να έχουμε μία και μόνη λύση. Θα πρέπει να δούμε από πολλές οπτικές γωνίες το θέμα ε, για να μπορέσουμε να ε, αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και επίσης δεν θα πρέπει οι χώρες να το παίζουν μοναχοί και καβαλάριδες γιατί όλοι μαζί θα πρέπει να βρούμε λύσεις. Ακούσαμε και το είπαν και οι συνεισηγήτριες ότι για θέματα ασύλου μετανάστευσης θα πρέπει να βασιστούμε στην συνεργασία. Ε, το πρόβλημα δεν οφείλεται και αναφέρεται εδώ ε, στην έκθεση, το πρόβλημα δεν οφείλεται σε ελλειπή νομοθέτηση, αλλά στο ότι δεν εφαρμόζεται καλά ε, και σωστά η νομοθεσία την οποία εδώ στο Κοινοβούλιο εκπονούμε και ε, ε, κυρίως είναι γεγονός ότι στο, όσον αφορά την πολιτική ασύλου αυτή η ελλειπής εφαρμογή της νομοθεσίας ε, καθίσταται πιο σοβαρή και πιο ε, προφανής. Επίσης ε, γίνεται λόγος ε, για ελλειπή αλληλεγγύη. αν δείτε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια θα διαπιστώσετε ότι τα κράτη-μέλη, όλα τα κράτη-μέλη έχουν ήδη ε, δείξει ελλειπή αλληλεγγύη και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε μαζί από κοινού να βρούμε λύσεις σε κοινά προβλήματα. Έτσι θα μπορέσουμε μόνο να φτάσουμε σε σωστές λύσεις. Και δεν νομίζω ότι το πρόβλημα έγκυται στον αριθμό των ε, μεταναστών. Το πρόβλημα έγκυται στην, ε, πραγματι... στην έλλειψη πραγματικής ευρωπαϊκής λύσης, πραγματικής ευρωπαϊκής προσέγγισης. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στα εξωτερικά σύνορα. Αναφέρεται διαρκώς ότι τα εξωτερικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα και μας ενδιαφέρουν όλους και είναι προς το συμφέρον όλων. Αλλά μόνο τα ε, κράτη μέλη τα οποία έχουν τέτοια εξωτερικά σύνορα προσπαθούν να λύσουν το πρόβλημα και έχουν, ε, ε, ε έχουν επικεντρώσει τις προσπαθειές τους ε, σε αυτά. Οι άλλοι που δεν έχουν, οι άλλες χώρες οι οποίες δεν έχουν εξωτερικά σύνορα δεν ασχολούνται πολύ με το θέμα. Αλλά όλοι θα πρέπει να προσπαθήσουμε από κοινού. Θα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίσουμε όλοι ότι όλα τα κράτη-μέλη κάποια στιγμή Ε, έχουν αμαρτήσει κατά κάποιο τρόπο λόγω έλλειψης ε, αλληλεγγύης. Το σλόγγαν μας θα πρέπει να είναι ενωμένοι στη στην διαφορά ή στη διαφοροποίηση. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα αλληλεγγύης ε, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταφέρει να παραμείνει ενωμένη ακόμα και σε δυσκολίες. Η έκθεση αυτή, ε, την οποία θα ξανασυζητήσουμε βεβαίως ε, ξανά και εν λεπτομερία, μας δείχνει ότι θα πρέπει σε, ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να δουλέψουμε. Και θα επιτύχουμε λύση με την προϋπόθεση όμως να υπάρξει η απαραίτητη πολιτική βούληση. Όσον αφορά τα εξωτερικά σύνορα θα συμφωνήσω ε, και θα στηρίξω αυτά που είπε ο κύριος Τιμ. Δηλαδή το πρόβλημα δεν είναι μόνο νομοθετικό ή οικονομικό. χρειάζεται πραγματική πολιτική βούληση χρειάζεται κοινή πολιτική έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Όσο δεν αφορά την συνεργασία με τρίτες χώρες, οπωσδήποτε θα πρέπει να έχουμε σαφή ορισμό, δηλαδή τι εννοούμε και τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία με τις τρίτες χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μόντσο. Ε, ευχαριστώ Κλοντ και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ ότι Ρομπέρτα περνάει τα γενέθλια της πολύ ωραία, τα καλύτερά της ε, γενέθλια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Κέγκια γιατί είναι πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Είναι τόσο περίπλοκο που αυτοί που κάνουν το πρώτο βήμα αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προσκόμματα. Τώρα ε, ρίξαμε αυτά τα προσκόμματα και έτσι μπορούμε να προβάλλουμε τις δικές μας ιδέες. Αλλά το πρώτο βήμα είναι και το ε, δυσκολότερο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ λοιπόν. Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την εργασία. Νομίζω ότι όλοι μπορούν να συνεισφέρουν αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την διάρθρωση της έκθεσης γιατί τώρα έχουμε ένα σκιαγράφημα από διάφορες οπτικές γωνίες. Για να έχουμε όμως μια ολιστική προσέγγιση θα πρέπει να έχουμε και μια πιο συστηματική προσέγγιση. Θα πρότεινα να δούμε τη στοχοθέτησή μας, τι θέλουμε να επιτύχουμε. Θέλουμε να αναθεωρήσουμε το σύστημα του Ουτουβλίνου, να το ξανακτήσουμε, να το κάνουμε λειτουργικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας. Υπάρχουν όμως και άλλα στοιχεία. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις που θα μας βοηθήσουν για, και για την αγορά εργασίας. Το δημογραφικό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ως προς τους πολιτικούς στόχους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τη ριζοσπαστικοποίηση και την ε, μεταναστευτική κρίση, αλλά να βρούμε και πολιτικές λύσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε το δημοκρατικό δυναμικό της Ευρώπης. Όταν ε, βλέπουμε αυτούς τους στόχους, θα μπορούσαμε να δούμε προς τα πού θα πρέπει να κινηθούμε, ποια είναι τα μέσα, ποιοι είναι οι φορείς. Να έχουμε μια συστημική προσέγγιση δηλαδή για να δούμε τα νέα στοιχεία που υπησέρχονται και να αφήσουμε κατά μέρος αυτά που ήδη προϋπάρχουν. Έχουμε και χρειαζόμαστε μάλλον ένα κοινό σύστημα ασύλου. Έχουμε μία έκθεση, επειδή είμαι σοσιαλδημοκράτης, δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για αλληλεγγύη, για μία ηθική υποχρέωση. Δηλαδή ε, υπάρχει συνταξιοδοτικό, υπάρχει ασφαλιστικό σε όλες τις χώρες. Δεν είναι θέμα ηθικής. Η Ευρώπη χρειάζεται ένα κοινό σύστημα αντιμετώπισης του προσφυγικού, προσφυγικού το οποίο να είναι θεσμικό, να έχει θεσμικό χαρακτήρα. Με απογοήτευσε πολύ η παρέμβαση του Συμβουλίου, γιατί όλοι μιλήσαμε για την ανάγκη να συμμετέχει και το Συμβούλιο ενεργά. Περιμέναμε από τη νέα Προεδρία να έχει και νέες ιδέες. Ελπίζω την επόμενη φορά όταν συναντηθούμε ε, με την Προεδρία να και από το Συμβούλιο. Μην το πάρετε προσωπικά, λέει ο Πρόεδρος προς τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Είναι θέμα εφαρμογής. Έχουμε ε, δύο ακόμα ομιλητές Κυρία Άλπη είναι εδώ. Α, εμένα προσφωνήσατε. Ευχαριστώ πολύ. Όχι πάνω από δύο λεπτά. Στον τύπο ε, πάντα εμφανίζονται ειδήσει για ναυάγια όπου πεθαίνουν ε, δεκάδες, εκατοντάδες άνθρωποι. Γίνονται ε, πολλές ανακοινώσεις, αλλά τίποτα δεν έχει αλλάξει ή κάτι έχει αλλάξει προς το χειρότερο. Γι' αυτό η μεταναστευτική πολιτική ε, δεν θα πρέπει να βασίζεται στην καταστολή. Μιλάμε για αλληλεγγύη έναντι των ε, μεταναστών, αλλά μιλάμε στην ουσία για επαναπατρισμούς και ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων. Αποτύχαμε απόλυτα ως προς τις πολιτικές της Επιτροπής. Γι' αυτό και είναι γελή η αριθμή ανάληψη μεταναστών. Εμείς δεχτήκαμε 17 ε, μετανάστες σε σχέση με τον αρχικό αριθμό των 17.000. Ε, Γι' αυτό θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα του Δουβλίνου, δηλαδή στο κέντρο των μελημάτων μας να είναι η συναπόφαση και η ίση κατανομή μεταξύ κρατών μελών και ιδιαίτερα να δεχόμαστε τους μετανάστες στις χώρες που υπάρχει η οικογένειά τους. Δυστυχώς ε, δεν υπάρχει τέτοια θέληση υπέρ των μεταναστών. Ακούμε ξενοφοβικές δηλώσεις από την τσεχική δημοκρατία που ανέφερε ότι οι μουσουλμάνοι ποτέ δεν ενσωματώνονται στην Ευρώπη και κανένας ε, δεν καταδίκασε το γεγονός ότι δεν αποδέχτηκαν το ανώτατο όριο που τους επιβλήθηκε. Τίποτα δεν ε, ε, αναφέρεται σαφώς. Αν μιλάμε για την εξωτερικοποίηση των συνόρων μας. Η Τουρκία δηλαδή αναλαμβάνει την βρώμικη δουλειά για μας. Επίσης θεωρούμε ότι σε περίπτωση διακίνησης θα πρέπει να σταματήσουμε με την στρατιωτικοποίηση της Μεσογείου. Θα υποβάλουμε τροπολογίες γιατί θα πρέπει να υπάρχει ε, αλληλεγγύη και όχι καταστολή στα ε, σύνορα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα πρώτα πρώτα συγχαρητήρια με όλους, για όλους όσους ασχολήθηκαν με αυτό το έγγραφο. Νομίζω το βούλιο στα σοβαρά να βγάλει τις ευθύνες του και όντως θα πρέπει να δούμε πώς θα αναθεωρήσουμε, πώς θα αλλάξουν το μηχανισμό του Δουβλίνου γιατί είναι αδύνατον ε, να, έχουμε θεσμική ελεγγύη παίρνει της ηθικής ελεγγύης Το Κοινοβούλιο αυτή τη φορά τι θα κάνει με αυτό το αξιόλογο υλικό. Δεν ξέρω. Θα καταφέρουμε επιτέλους το Συμβούλιο να παίρνει στα σοβαρά τη δική του υπευθυνότητα αυτήν που πέρσι δεν ανέλαβε. Εδώ υπάρχουν αξιολογικές προτάσεις και μπορούμε να τις ε, βελτιώσουμε. Και θα πρέπει να υπάρχει βούληση από τα κράτη, αλλιώς θα αποτύχουμε παταγωτός. Ο πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ας αφήσουμε λίγα λεπτά για να μπορέσουν να δευτερολογήσουν οι συγητέ. Ρομπέρτα Ευχαριστώ όλους τους άνθρωπου που ήρθαν εδώ να ακούσουν τις εισηγήσεις μας και που ήρθαν για να μας ε, πούν ε, τις ε, πρώτες του σκέψεις περιμένω πως και πως τις ε, δροπολογίες τώρα διευκρινιστικά όταν μιλάμε για χρονοδιάγραμμα για το άσυλο το διευκρινίζω ότι πρόκειται για κάποιο μεγάλο που ήδη υπάρχει όσον αφορά την οδηγία για την υποδοχή και υπάρχουν και κάποιοι περιορισμοί σε σχέση με το τι μπορούμε να κάνουμε όταν ήδη υπάρχει κάποια διαδικασία που είναι εφαρμοστέα και άρα θα πρέπει όλοι να την εφαρμόσουν και ιδίω όσον αφορά την πρόσβαση σε όλους ε, άσυλο και πρόσφυγες στην απασχόληση. Η κυρία Στέιφενς και ο κύριος Κέρκο ε, μας μίλησαν για το ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με κάποιο είδους ε, μέθοδο à la carte για αυτούς οι οποίοι ζητούν κάποια προστασία. Δηλαδή να μπορούν να επιλέξουν την χώρα που τους παράσχει την προστασία. Μα ε, το διατυπώσαμε με έναν τέτοιο τρόπο και προσπαθούμε να δώσουμε μια συνέχεια στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από μερικού μήνε. Άρα θα πρέπει να δούμε πώ θα καλύψουμε βέβαια ε, τι επιθυμίε των, τον Αλλά αυτό δεν είναι δυνατόν να λιώσει τη διαδικασία της κατάσταση Μιλάμε για να που υπάρχουν στην πράξη και όχι για κάποιες διατάξεις που θα περιορίσουν νομοθετικά τα κρατημέλη και το Συμβούλιο ακόμα περισσότερο. Η άλλη εισηγήτρια κύριε Γκέγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους οι οποίοι έλαβαν τον λόγο. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και το Συμβούλιο. Είναι σημαντικό πιστεύω να προσεγγίσουμε τη μαστευτική πολιτική με σλόγγαν. Θα ήταν εύκολο αυτό, με συνθήματα. Και επομένω κανεί με εφευρετικότητα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο. Αλλά δεν είναι αυτό το πνεύμα που διαπνέει την έκθεσή μα. Ο στόχο μα είναι να έχουμε μια έκθεση ε, με προσέγγιση εμβρηθή, ο σφαιρική και εντελεχώς να εξετάζουμε διάφορα θέματα. Καταλαβαίνω ποιες είναι οι δυσκολίες που επισημαίνει η κυρία Στέφενς, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία και εμείς που είπε και τα θίγουμε και εμείς. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλο το υλικό που ήδη υπάρχει μέχρι σήμερα και κυρία Σπινέλη σε αυτό που είπατε για την λαθρέα διακίνηση αλλά και για την εγκληματική δραστηριότητα ότι και αυτό θα είναι σημαντικό σημείο στο κείμενο και επίσης ο κύριος Φοντάν είπε για επαναπατρισμούς και είπε ότι θα πρέπει να τηρηθεί το διεθνές και το ευρωπαϊκό για την ε, οικονομική μετανάστευση. Τα κράτη-μέλη διατηρούν τις εθνικές αρμοδιότητες για να επισημάνουν τι να τι θέσεις υπάρχουν κενές στην αγορά εργασίας. Άκουσε και τον συνάδελφο Αγγιλάρ Λόπες ότι θα πρέπει να ε, αλλάξει πολύ τον κρατών αλλά και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να σας τονίσω κάτι που είπε η κυρία Μουσολίνη εμείς δεν λέμε ότι θα πρέπει τα μετανάστες να βρουν δουλειά σε νέα μήνες. Παραπέμπουμε σε κάποια οδηγία που έχει εγκρίνει ε, το 2013 Συμβούλιο και Κοινοβουλίο άρθρο 15. Ορίζεται ότι τα κράτη-μέλη προσφέρουν εγγυήσεις για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτό δεν πάει να πει ότι κανείς θα έχει δουλειά μέσα σε 9 μήνες από τότε που θα υποβάλει ε, αίτηση για διεθνή προστασία. Εν κατακλείδη σας αναφέρω κάτι που για είναι σημαντικό. ότι δεν θα πρέπει να, να, να, να μην να, δεν θα πρέπει να χάνουμε το, το στόχο μας. Θα πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται στην πραγματικότητα και θα πρέπει επίσης να μην έχουμε χειραγώγηση αυτών των φαινομένων που γίνονται εις βάρος των ε, γυναικών και κανείς να μην εκμεταλλεύεται από την άλλη μεριά αυτά τα γεγονότα. Ο Πρόεδρος. Ζητώ συγγνώμη από αυτούς που δεν έλαβαν το λόγο. Θα γίνει την επόμενη φορά. Στο 8 Φεβρουαρίου θα πρέπει να υποβληθούν οι τροπολογίες μέχρι τις 8 το βράδυ και να δούμε σε ποια κατεύθυνση θα κινηθούμε και ιδιαίτερα για αυτούς που δεν ε, διάβασαν ε, ενδελεχώς το κείμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας συνάδελφοι. Η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 25 Ιανουαρίου. Ε, στα διάφορα υπάρχει κάτι. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.